60 μοίρων. Τα πρακτικά της ε, συνεδρίας της 17, 17 Ιουλίου έχουν διατεθεί στους βουλευτές. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι.